Και τώρα έχουμε τις εκθέσεις Λεγκρίπ και Αρενά, προτεραιότητες για την 61η Σύνοδο της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων για τη θέση της γυναίκας. Αντί της κυρίας Λεγκρίπ θα δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά στην κυρία Κοράτσα Μπίλτα. Παρακαλώ. Commissioner... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Έχω την δυνατότητα να απευθυνθώ στους συναδελφούς και με περήφανη για αυτό και να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε για την 61η Σύνοδο τη Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση τη γυναίκα, που μα δίνει μια ευκαιρία να ενώσουμε τη φωνή μας με εκείνους που παλεύουν για την αξιοπρέπεια της γυναίκας παγκοσμίω, να καταπολεμήσουμε τις, τα, στερεότυπα και τις διακρίσεις πέρα από τη ρητορική και να περάσουμε στις πράξεις, γιατί χρειάζονται πράξεις παντού και πολύ περισσότερα να γίνουν για να οδηγηθούμε σε ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Πρέπει να δώσουμε μια φωνή σε αυτά τα εκατομμύρια γυναικών που παραμένουν περιθωριοποιημένες και που δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Είναι γυναίκες πρόσφυγες, είναι γυναίκες με αναπηρία και πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών ε, χωρίς καμία ανοχή στην ε, οικογενειακή βία, στο τράφικινγκ, στην σεξουαλική εκμετάλλευση, τον ακροτηριασμό γενικών γενετικών οργάνων, τους εξαναγκωστικούς γάμους κτλ. Πολλές γυναίκες είναι οι σκλάβοι της, της σύγχρονης εποχής Έχουμε ακούσει εκατοντάδες χιλιάδες δραματικές ιστορίες. Ζητούμε την πλήρη επικύρωση του Συμφώνου της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προστατεύεται αυτή. Να ενισχύσουμε τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες είναι πολύτιμο ε, στοιχείο για την αναοικονομική μας ανάπτυξη και να φροντίσουμε για την ισότιμη ε, την, ε, την ίση αμοιβή για ίση εργασία να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής και να δοθεί πλήρης πρόσβαση στην υγειονομική περίθελψη για τις γυναίκες και τα κορίτσια συμπεριλαμβανομένων των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων η σύνοδος, η 21η σύνοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε και να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη παγκόσμια η οποία έχει, αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Τώρα που οι Ηνωμένε Πολιτείε απεμπολούν, τον ευθυνών, απεμπολούν τις ευθύνες τους, τώρα θα πρέπει η Ευρώπη να ανανεώσει την υποστήριξή της στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών στη διεθνή συνεργασία. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε, η νέα του κυβέρνηση φαίνεται ότι γυρνάει την πλάτη τη στις, στα δικαιώματα των γυναικών. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε η, η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, δείχνει την πρόθεσή της να υλοποιήσει ακόμα πιο αυστηρά τον κανόνα του Global Gag Rule, δηλαδή τη μη χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, προγραμμάτων ε, σεξουαλικής υγείας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αυτό το και να καλύψει αυτό το κενό σε προγράμματα στην Αφρική, στην Ασία έχουν απευθυνθεί πολλές εκκλήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτές α, τις γυναίκες. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στις εθνικές μας κυβερνήσεις, έτσι ώστε να βρεθούν κονδύλια τα οποία θα καλύψουν το κενό που θα αφήσουν πίσω τις ΗΠΑ. Και να καλέσουμε και άλλες κυβερνήσεις και άλλες ε, οργανώσεις να ε, συνεργαστούν σε προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, γιατί οι επιπτώσεις αυτού του λεγόμενου gag rule είναι πολύ σοβαρές. Σε όλους τους τομείς, στην περιενετική περίθαλψη, στην καταπολέμηση της παιδικής θνησιμότητας, στην υγειονομική περίθαλψη τους ώστε να μην πεθαίνουν γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτόν τον σεξισμό, αυτόν τον, την, την, την, την φιλοσοφία του Τραμπ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία έχει Το λόγο για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η, η τέταρτη σύνοδος που οργανώθηκε το 1900 95 στο Πεκίνο για τις γυναίκες πραγματικά σηματοδότησε μια πάρα πολύ σημαντική ε, Επιτροπή όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Εγκρίθηκε τότε ένα πρόγραμμα δράση για την χειραφέτηση, την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, πράγμα το οποίο αποτέλεσε το σημαντικότερο πολιτικό έγγραφο για την ισότητα ανδρών και γυναικών τα τελευταία 20 χρόνια. Η Σύνοδο του Πεκίνου Συνήκωση το 2015 χαιρέτησε την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον τομέα αυτό χάρη σε αυτό το παγκόσμιο μέσο. Ωστόσο, είχαμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να κάνουν αξιολογήσεις και τους είχαμε ζητήσει να κάνουν νέες μετρήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μέσων αυτών για την διασφάλιση της ισότητος. Και παρόλα αυτά, το 2017, εν έτη 2017, βλέπουμε ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και τα δικαιώματα των γυναικών, τίθενται να αμφιβόλω εκ νέου. Στο σημερινό κόσμο βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν ε, πολιτικές οι οποίες δεν υποστηρίζουν πραγματικά τα δικαιώματα των γυναικών ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε γενικότερα στην ΟΜΕΝΕΘΝΗ. Απέναντι λοιπόν στην οπισθοδρόμηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι υπάρχει η κοινωνία των πολιτών η οποία οργανώνεται και αντιστέκεται. Κατά την 61η Σύνοδο τη Επιτροπή του ΙΕ για τη θέση τη γυναίκα, εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούμε από το Συμβούλιο να αναλάβει τι απαραίτητε πρωτοβουλίε προκειμένου να ηγηθεί υπέρ τη ισότητα των ανδρών και γυναικών στα πλαίσια του διεθνού κοινότητο, όπω το είχε κάνει πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να προωθήσει ουσιαστικά την εκπαίδευση και την παιδεία και να φτάσει μέχρι την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών με την έγκριση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Θα πρέπει να υπάρχει καθολική επίση πρόσβαση σε, σε όλου του τομεί τη υγεία συμπεριλαμβανομένη τη αναπαραγωγική υγεία και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία θα πρέπει να γίνεται χωρί καμία διάκριση και οι γυναίκε θα πρέπει να συμμετέχουν επίση στην κοινωνική και πολιτική ζωή των χωρών του, ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χειραφέτησή του. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή που έχει φτάσει πλέον η 61η Σύνοδο Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση τη γυναίκα, δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε την κυβέρνηση Τραμπ που αποφάσισε να καταργήσει τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπω είπε και η συνάδελφό μου Κοράτσα Μπίλτα μη κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίε ε, συμβάλλουν πάρα πολύ στον οικογενειακό προγραμματισμό και επίση όλο και λιγότερε γυναίκε πλέον στι ΗΠΑ θα έχουν πρόσβαση στι ε, υπηρεσίε οικογενειακού προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την καταπολέμηση του AIDS, για τη γενικότερη κατάσταση τη γυναίκα, για την υγεία των ίδιων των παιδιών. Η στάση αυτή τη κυβέρνηση Τραμπ θα έχει δυσμενεί συνέπειε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε τη στάση της κυβέρνησης ε, Τράμπα, καθότι αυτή προωθεί πέρα από τον οικονομικό προστατευτισμό και πολλές άλλες πολιτικές. Για τον οικονομικό προστατευτισμό όμως όλοι ανθίστανται και λένε τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Για ποιο λόγο όμω σιωπούμε όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Και στον τομέα λοιπόν αυτό, κυρίε και κύριοι, όταν μιλάμε για, γυναικο... για δικαιώματα των γυναικών και επομένω για ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να αποδοκιμάζουμε και να κατακρίνουμε τόσα όσα κάνει η κυβέρνηση Τραμπ. Πρέπει να το πούμε αυτό προ τι ΗΠΑ και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα αυτού που θα πρέπει να δοθεί υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία είναι προφανώ ανθρώπινα δικαιώματα και μην ξεχνάμε ότι το ίμιση τη ανθρωπότητα είναι γυναίκε. Σα καλώ λοιπόν να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ το Συμβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στη δικασία Catch the Eye. Τσάβα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Θα είμαι πολύ αυστηρή με το χρόνο ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες δεν έχουν ευκαιρίες για οικονομική ανεξαρτησία και χειραφέτηση ούτε ελέγχουν ε, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων που μπορεί να καθορίζει τη ζωή τους. Ιδίως στη σημερινή εποχή και όταν βλέπουμε τι κάνει ο ηγέτης ε, της πιο δημοκρατικής ε, χώρας, επίσης βλέπουμε την υπεκπροσώπηση των γυναικών. παρόλα αυτά αυτό που πρέπει να του εξασφαλίσουμε είναι η δίκαιη μεταχείριση, η ισότιμη μεταχείριση. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει την κατάργηση, ακύρωση οποιασδήποτε αρνητικής για τις γυναίκες νομοθεσίας, οποιαδήποτε χώρα. Αυτό είναι σημαντικό και για τις χώρες μας αλλά και για τα. κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2017 κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασικό θεμέλιο για ένα ειρηνικό, ευημερούντα και βιώσιμο κόσμο. Η πρόοδος είναι αργή και άνηση. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά και μορφές διακρίσεων παρά τις βάσιμες ενδείξεις ότι η χειραφέτηση των γυναικών έχει σημαντική πρόοδο οδηγήσει στη μείωση της φτώχειας στην πρόθεση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. επιπλέον η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα σε παγκόσμια κλίμακα και η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικό επίπεδο συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμω όταν μια οικονομία πλήττεται οι πρώτες που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι γυναίκες. στην ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των γυναικών φτάνει στο. 27,7%. οι γυναίκες αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που έχει πληγεί περισσότερο από την πολιτική λιτότητα στην ελλάδα. η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να λάβει μέτρα για να σταματήσουν τα στερεότυπα κατά των γυναικών. ευχαριστώ. Ναι, με ακούτε. Is there a problem with... Υπάρχει ένα πρόβλημα, μήπως, με τη γερμανική καμπίνα φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Να ενημερωθεί η κυρία Ρέντκε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί αγαπητέ Κυρία Επίτροπε, και στο ΟΒΑΛ γραφείο και αλλού κάποιοι θέλουν να μας ε, κουράσουν, να σταματήσουμε να μιλάμε και να σταματήσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, ε, τα δικαιώματα για το σώμα μας. Δεν θα το κλείσουμε όμως, δεν θα το βουλώσουμε, δεν θα, ξεχα... δεν θα κουραστούμε και δεν θα σταματήσουμε να παρασφίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών γιατί είναι θεμελιώδη δικαιώματα και όσο περισσότερο τέτοιοι άνθρωποι μας πιέζουν, όσο περισσότερο ενωμένε θα είμαστε, όχι εδώ μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και στους δρόμους, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και δεν, θα είμαστε μόνο ενωμένε, αλλά θα απαιτήσουμε και συγκεκριμένε δράσει από τι κυβερνήσει μα, ε, που θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Γι' αυτό λοιπόν απαιτώ από τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει ε, να ε, προσχωρήσουν στην Ολλανδική, Βελγική, Δανική και Σουηδική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού του Golden Gap Rule. Όχι, απλά δεν έχουμε κουραστεί. Μόλις ξεκινήσαμε. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σεντρόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται πολύ καλέ συστάσει για τη βελτίωση τη κατάσταση των γυναικών, ε, τη οικονομική του των δικαιωμάτων του ε, και μέτρα για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Δυστυχώ όμω οι γυναίκε εξακολουθούν να είναι θύματα ε, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στο θέμα της παροχής ασύλου Βλέπουμε σε πολλά κράτη ε, το πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, παραδείγματο χάρη για το διακανονισμό συγκρούσεων, για την επίλυση διαφορών και όσο πιο πολλές γυναίκες είναι στα πολιτικά ή στα άλλα υψηλά αξιώματα τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να υπάρχει μεταξύ άλλων ε, προστασία των δικαιωμάτων, προστασία των αναπαραγωγικών σεξουαλικών δικαιωμάτων. Δεν είναι σωστό να μιλάμε βέβαια μόνο ε, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και την καταπολέμησή του. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι άντρες φαίνεται να είναι περισσότεροι, αλλά το ζήτημα αυτό εμένα με αφορά όλους ιδιαιτέρως. Εργαστήκαμε πάρα πολύ για την ε, πρόθεση και την βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Συμφωνώ απόλυτα ότι όλες οι γυναίκες και όλα τα κορίτσια θα πρέπει να έχουν τις ίδιες και ίσες ευκαιρίες, είτε πρόκειται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, είτε πρόκειται για την ισότιμη αμοιβή. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο σε όλου του κλάδου και στο γεωργικό κλάδο. Οι γυναίκε αποτελούν έναν πολύτιμο κρίκο τη αλυσίδα, τη οικονομική σε πάρα πολλού παραγωγικού τομεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δεχθούμε την τροπολογία εκείνη που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει την άμβλωση με κοινοτικά κονδύλια. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα βελτιωθεί η θέση της γυναίκας με τα μέτρα αυτά. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ισότιμη μεταρρύθμιση μεταξύ ανδρών και γυναικών.